say that the votes will take place at 4 o'clock. Good afternoon everybody. May I have attention please. Καλό σας απόγευμα. Παρακαλώ, ακούστε με. Καταρχάς, καλώς ήρθατε όλοι στις Βρυξέλλες. Όσοι ήρθαν πίσω μετά από ένα ζεστό καλοκαίρι πιστεύω να ανακουφιστούν με έναν πιο ή πιο πιο δροσερό καιρό εδώ και ελπίζω όλοι να είχατε πολύ καλές διακοπές. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να εργαστούμε. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Έχουμε εδώ την ημερήσια διάταξη, το σχέδιο ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσει, όχι, εντάξει, εγκρίνεται ω έχει. Πρακτικά των προηγουμένων συνεδριάσεων 20-21 Ιουνίου και 11-12 Ιουλίου. Θα θεωρηθούν ω συνήθω κάνουμε εγκεκριμένα, δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, ωραία. Εν συνεχεία, ανακοινώσει του Εν συνεχεία, σύμφωνα με αυτά που κάνουμε, ε, το, η συνεδρίαση αυτή προβάλλεται στο διαδίκτυο και όσοι ενδιαφέρονται μπορεί να έχουν και τις, ε, την μίση διάταξη της γλώσσα τους. Τέσσερα, Η πρόοδος των τριμερών διαπραγματεύσεων. Το τελευταίο που είχαμε πει είναι, συζητήσαμε τα εξαιρετικά μέτρα, τα προτιμησιακά μέτρα για το Πακιστάν και το κείμενο υιοθετήθηκε στις 18 Ιουλίου. Τον Ιούλιο το συζητήσαμε και ελπίζω στην επόμενη συνεδρίαση. Τώρα, Omnibus 1 και 2 αναμένουμε τις αντιδράσεις, τις απαντήσεις του Συμβουλίου. Ε, για να δούμε... Α, εάν δεν κάνω λάθος, λέει ο πρόεδρος, το Μάιο, το Μάιο υιοθέτησαν τις θέσεις του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο λοιπόν ε, καθυστερεί υπερβολικά, πιστεύω, στην, ε, στην απάντησή του, στην ανταπόκρισή του διότι αυτό αφορά τις, ε, νομο, τις συμφωνίες νομοθετικής φύσεως σε βάση της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχει επιπτώσεις δηλαδή στο νομοθετικό κεκτημένο και πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο να απαντήσει. Δεν υπάρχει λόγος ε, για την καθυστέρηση αυτή. Έχουμε αρχίσει άτυπες συναντήσεις για τις εμπορικές συμφωνίες με την Κεντρική Αμερική. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα και γι' αυτό ο τριμερής διάλογος δεν μπορεί ακόμα να αρχίσει. Αλλά έχουμε αρχίσει προκαταρκτικές επαφές. Τώρα, ε, χρηματοδότηση, σημείο 5, των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων των μικρομεσαίων. Έχουμε μία έκθεση από την αδελφή επιτροπή μας. Ο εισηγητής είναι ο Γιάννη Ζαχραντήλ. Αλλά δεν είναι εδώ. Ε, μας έχει στείλει τους λόγους της απουσίας του και για αυτό θα αντικατασταθεί από τον ε, Well, first of all, Mr. Zaradil sends his deepest apologies. Uh, he's caught up with family Καταρχάς ο κύριος Ζαχράντη είχε εικονιακά προβλήματα και δεν μπόρεσε να έρθει και γι' αυτό μου έδωσε μένα ε, την έκθεσή του. Καταρχάς, η σημασία των μικρομεσαίων επιχείρησεων είναι τεράστια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το 99% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σύμφωνα με την, τις αξιολογήσεις της έρευνες της Κομισιόν υπάρχουν 23 εκατομμύρια τα οποία προσφέρουν τα 2 τρίτα των ε, θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού όγκου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να είναι σωστή και θεμητή στα νέα μας προγράμματα και στη νέα πολιτική. Είναι η, η αδυναμία εξέβρεσης κεφαλαίων κινήσεων είναι το βασικό πρόβλημα και για να διορθώσουμε αυτή την έλλειψη ο εισηγητής προτείνει μεταξύ των άλλων να κάνουμε τα εξής. Πρώτον, να απλοποιήσουμε σε εθνικό επίπεδο την ε, πρόσβαση σε πληροφορίες, να αυξήσουμε τις διαβουλεύσεις με τις διάφορες συναρμόδιες επιτροπές και οργανώσεις και τον ε, οικονομικό τομέα. Ε, να διευκολύνουμε δηλαδή την μείωση της γραφειοκρατίας και τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερον, να υιοθετήσουμε μονάδες υποστήριξης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα επικεντρώνονται στην υποστήριξη και βοήθεια ε, σε εθνικό επίπεδο και στην ε, γλώσσα τους και ε, να βοηθούν σε ό,τι χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενημέρωση σε νέους κανονισμούς, υπέρβαση των εμποδίων και των προσκομμάτων στο διεθνές συμπόριο, διευκόλυνση διασυνοριακών συναλλαγών και επίσης πρόσβαση σε ανταγωνιστικές αγορές τρίτων χωρών. Τρίτον, η Κομισιόν να διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην εδραίωση διεθνών προτύπων. Δεδομένου ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον αλλάζει συνέχεια, αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στην κερδοφορία. Τέταρτον, να μπορέσει να εκμεταλλευτούν όλες τις επενδυτικές δυνατότητες οι οποίες προκύπτουν από τις διεθνείς ε, συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών και τις ε, ε, συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμφωνίες για την μεσογειακή εταιρική συνεργασία και άλλες συναφείς. Εν συνεχεία, να δημιουργήσουν συνέργειες να αναπτύξουν συνέργειες για να αναβαθμιστούν περαιτέρω, περαιτέρω οι διπλωματικές υπηρεσίες με τους εμπορικούς ακολούθους λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή του εισηγητού. Η κυρία Θαμόρα από τους ε, σκιώδη ηγητές εκ μέρους του ΕΛΚ. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι Ευελπιστώ ότι θα μεταφραστεί τις επόμενες μέρες η έκθεση, γιατί προς το παρόν υπάρχει μόνο στα αγγλικά και έτσι και ο σχολιασμός μας θα είναι κάπως περιορισμένος. Καταρχήν, συμφωνώ με την τοποθέτηση του εισηγητού ό,τι αφορά την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πληροφόρηση και στο κεφάλαιο. Θεωρώ ότι η έκθεσή του είναι αρκετά πλήρης. Ίσως θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο γεγονός ότι οποιαδήποτε δράση που διεκπεραιώνεται ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι συμπληρωματική με αυτές που υπάρχουν και να προσφέρει προστιθέμενη αξία για να αποφύγουμε περί τη επικάλυψη με υπάρχοντα προγράμματα σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό επίπεδο. Όπως προτείνει ο συγγητής μας, αυτό που θα μπορούσε να περιληφθεί στο άρθρο 1-2 με μια ανάλυση κόστους-οφέλους που μάλιστα θα πρέπει να γίνεται τακτικά. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου οι, η μη δεσμολογικοί φραγμοί τη χάνουν μεταχείριση μεταχείρισης ε, και τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους δασμολογικούς φραγμούς. Είναι σημαντική η ασφάλεια δικαίου για τις επενδύσεις μας στην Αλλοδαπή. Και είναι δύσκολη η εξωτερήκευση, η διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Γι' αυτό και απαιτείται ασφάλεια δικαίου για τι επενδύσει του. Αν δεν υπάρχει τέτοια ασφάλεια δικαίου, είναι πολύ πιο αποθαρρυντικό για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει να ανοιχτούν ε, στη διεθνή αγορά. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση με του εμπορικού τη εταίρου θα πρέπει να εξασφαλίσουν αυτήν την ασφάλεια δικαίου για τι επενδύσει της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Ευχαριστώ τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δράσεις στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ευχαριστώ και τον εισηγητή μα για την μεστή και πλήρη έκθεση που μα παρουσίασε. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο σκιώδη εισηγητή. Α περάσουμε τώρα στα μέλη τη Επιτροπή. Α, συγγνώμη. Η Αμέλεια. Α, ναι, είμαι μικρή και δεν Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να υποβάλω και τη θέση των πρασίνων. Η πράσινη είναι αρκετά επιφυλακτική ως προς την ε, ιδέα ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα πρέπει οπωσδήποτε να διεθνοποιήσουν, να δώσουν ένα πιο διεθνή χαρακτήρα στι δραστηριότητε του, γιατί μια τέτοια δραστηριότητα είναι δαπανηρή και απορροφά ανθρώπινου πόρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στην ανάπτυξη πόρων και υπηρεσιών που θα είναι προσαρμοσμένε στι ε, τοπικέ συνθήκε και τι εθνικέ συνθήκε. Μπορεί βέβαια να θέλουμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς ε, θεμητού Έχουμε πρόσφατη έκθεση του κυρίου Βίγκλερ για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί αναφέρεται ότι είναι σημαντικό για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να διεθνοποιήσουν τι εργασίε του είναι να τι ε, προστατεύσουμε αποτελεσματικά από αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ εμπορικών εταίρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ε, έχουμε κάποιε ανησυχίε για θέματα εμπορίου σε ό,τι αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί εκεί μερικές φορές έχουμε ε, ε, απρόβλεπτα ασφαλιστικά μέτρα και προβλήματα με, τους, ε, με τις τελωνιακές διαδικασίες και δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση. Καλό θα ήταν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει μια αξιολόγηση για το πώ οι ευρωπαϊκέ μικρομεσαίε επιχειρήσει που θέλουν να εγκατασταθούν ή να αποκτήσουν αμερίδο σε ξένες αγορέ τι δυνατότητε έχουν σε περίπτωση που υπάρχει μία αξίωση και τι δυνατότητε ασφαλιστικών μέτρων υπάρχουν ε, ε, για τις εταιρείε αυτές. Είναι πολύ σημαντικό για τα θέματα ενημέρωσης και επικοινωνία, γιατί όταν μια μικρομεσαία επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ένωση προσπαθεί να εγκατασταθεί σε αμερικανική αγορά, εκτίθεται σε μηνύσει και αγωγέ ε, από αμερικανικέ εταιρείε εξαιτία των διαφορετικών διατάξεων που ισχύουν για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και την πνευματική ιδιοκτησία. Και μάλιστα επειδή οι αγωγέ είναι πολύ δαπανηρέ, μερικέ φορέ για να τι αποφύγουν οι εταιρείε ζητούν άδειε που μερικέ φορέ μπορεί να μην τι χρειάζονται. Είναι σημαντικό λοιπόν να προστατεύουμε τι δικέ μα μικρομεσαίε επιχειρήσει για να ε, μην γίνουν έρμεα κάποιοι που καταχρώνται Τη διατάξη πνευματική ιδιοκτησία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και σα ζητώ συγγνώμη που δεν σας πρόσεξα προηγουμένως. Τώρα ο κύριο Αρή Βέμπερ από τους Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ. Συνεχίζοντα τι προλαλήσει, τις, τις μάλλον, θα ήθελα να πω ότι ήμουν μακρόν μέλος της αντιπροσωπής για τις σχέσεις με, με την Κίνα και ε, πολύ συχνά στις συναντήσεις με εμπορικό και οικονομικό επιμελητήριο της Κίνας συνάντησα εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί σε τέτοιου είδου ε, σώματα δεν έχουμε εθνικές πάντα έχουμε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι θύματα αυτής της παραποίησης των ε, απομιμήσεων και του σφετερισμού ή της ε, καπήλευσης τη ε, πνευματική ιδιοκτησίας και των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Και ενώ οι μεγάλες εταιρείε, οι πολυεθνικές μπορούν να προσφύγουν σε αυτές τις δαπανηρέ, πολύ δαπανηρέ συχνά διαδικασίες στα πλαίσια της ΠΟΕ, γιατί έχουν τέτοια οικονομικά μέσα και νομικά μέσα, έχουν και ανθρώπινου πόρου. Αλλά μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το νομικό οπλοστάσιο που προσφέρει η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορία γιατί δεν έχει μέσα ούτε οικονομικά, ούτε νομικά, ούτε τους ανθρώπινου πόρους. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσθέσουμε και αυτό το σημείο και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε κάποιες διαδικασίες ε, για να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να προχωρήσουν ε, στην κατάκτηση των αγορών. Ευχαριστώ κύριο Σόλτς από την ΚΟΕ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του Σκιώδους, διότι για πολιτικούς λόγους βρίσκεται στην Ιρλανδία και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Οπωσδήποτε, αναμφίβολα, πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά με βάση και τα σχόλια των συναδέλφων γιατί μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές. Είναι ε, μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Ο Πολ θα ήθελε να καλύψει ορισμένα επιμέρους ζητήματα που δεν έχουν φύγει οι ΜΜΕ ε, υφίστανται τις συνέπειες της ύφεσης, που δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άλλα μέρη της υφηλίου. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με παγκόσμιες προκλήσεις και θα πρέπει να δούμε πώς οι ΜΜΕ μπορούν να ε, εκπονήσουν τη δική τους στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη. Οι ΜΜΕ είναι μία από τις βασικές ε, κινητήριους δυνάμεις ε, και για την ε, ανάπτυξη και για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να σταθεροποιήσουμε αυτή την κατάσταση σε μία περίοδο ύφεσης. Θέλει λοιπόν να τονίσει ο σκιώδης μας ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα πλαίσιο πιστώσεων, αλλά να δούμε πώς η παρακμή στις εγχώριες αγορές θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια αναπτυξιακή πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην λέμε ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία των μεγάλων επιχειρήσεων στα πλαίσια των ε, τρίτων αγορών. Το, μέλος, το μέλλον συγγνώμη, το ΜΜΕ ε, εξαρτάται από τις εγχώριες αγορές. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διεθνικοποίηση της ε, κρίσης αυτής. Είναι παγκόσμια η κρίση ή όχι. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προβούμε σε μία αναδιαμόρφωση και ένα νέο ορισμό της κατάστασης. Μιλάμε λοιπόν για τις ΜΜΕ που θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ε, ροής χρημάτων, κεφαλαίων, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσον εξαγωγών-εισαγωγών, ενώ στην παράγραφο 7 μιλάμε για οργανισμούς ε, ε, οργανισμούς εξαγωγών ή που υποβοηθούν τη διαδικασία εξαγωγών και ελέγχθη ότι θα πρέπει να δούμε πώς οι τράπεζες θα μπορούσαν να ασχοληθούν με, τους, ε, με τον ισοσκελισμό των προϋπολογισμών έτσι ώστε να μην υπάρχει ε, μεγάλη ροή δανειοδότησης αποκλειστικά. Θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή περαιτέρω και θα υποβάλουμε νέες προτάσεις έτσι ώστε αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας να είναι άκρος ενδιαφέρουσα για ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε. Πολύ σημαντική τα όσα αναφέρατε. Είμαι σίγουρος ότι ο συγγετής θα τα λάβει σαφώς υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει κάτι να μας πει ο κύριος Λιμανίδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή καλωσορίζει αυτή την έκθεση η οποία ε, υποβλήθηκε μέσα σε σωστά πλαίσια χρονισμού. Συμφωνούμε με την ανάλυση και την ιεράρχηση των θεμάτων όπως παρουσιάζονται η διεθνοποίηση είναι μία πρόκληση για τα ΜΜΕ, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλα προσκόμματα και το κυριότερο είναι η έλλειψη κεφαλαίων. Ως προς τις εμπορικές συμβάσεις και τις σχετικές πληροφορίες περί αγορών, το θέμα αυτό είναι ένα ισχυρό ζήτημα και αφορά της ΜΜΕ και όχι τις μεγάλες ε, πολυεθνικές. Ξέρουμε ότι η διεθνοποίηση των ΜΜΕ ε, θέτει ένα πλαίσιο ε, εξωστρέφειας της αγοράς. Γι' αυτό η διεθνοποίηση είναι μια βασική πολιτική. Μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις σε ένα μεγάλο κόσμο και το πρόγραμμα πλαίσιο κόσμε αυτό ακριβώς καταδεικνύει. Η παρούσα πρόταση αποτελεί ενθάρρυνση για την Επιτροπή να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση. Θα μελετήσουμε προσεκτικά τις συστάσεις και θα τις λάβουμε υπόψη μέσα στα πλαίσια της μελλοντικής μας πολιτικής για την εφαρμογή του νέου προγράμματος πλαισίου για τις ΜΜΕ και την ανταγωνιστικότητα. Ε, αναμένουμε την έγκριση αυτή της έκθεση με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελε κάτι να μας πει ο εισήγητής. Θα μιλήσω λίγο πιο ελεύθερα Νομίζω ότι και οι τέσσερις ε, ομιλητές είχαν να συνεισφέρουν ουσιαστικά. Και νομίζω ότι ένας από τους ομιλητές ήταν και επικεφαλής μιας ΜΜΕ. Έχει μεγάλη σημασία η προσβασιμότητα στη χρηματοδότηση, γιατί είναι κάτι το πολύ δύσκολο για τις ΜΜΕ. Αυτά τα σημεία βεβαίως θα ληφθούν υπόψη από τον εισηγητή και γνωρίζουμε ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για το μέλλον της Ευρώπης. Διαφορετικά δεν υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης Μιλάμε για 23 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν την μεγάλη σημασία τους. Ευχαριστώ πολύ. Άρα λίγη συζήτηση επί του ε, θέματος αυτό. Στις 27 Σεπτεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν είναι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Σημείο 6 ενδιάμεση έκθεση εν ώψη της θετικής έκβασης της διαδικασίας έγκρισης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Είναι μία γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προϋπολογισμού, η οποία είναι η Επιτροπή επί της ουσίας και η συγητή της δικής μας γνωμοδότησης είναι ο Σάιαντ Κάμαρ. Και στο φάκελό σας, στον ντοσιέ σας, έχετε την, το σχέδιο γνωμοδότησης. Ο κύριος Καμάλ ε, έχει αιτιολογήσει την απουσία του και θα αντικατασταθεί από τον Ρόμπερτ Στέρντι, και του δίνω και πάλι το λόγο. Αυτό συμβαίνει. <laughs> Αυτό συμβαίνει, πρόεδρε, όταν συντονίζεις, είσαι συντονιστής μιας μικρής ομάδας και πάλι ο Σάιετ στέλνει την... λύπάτη ιδιαίτερα που δεν είναι εδώ και θα αναλάβω εγώ την παρουσίαση του, ε, της ενδιάμεσης έκθεσης. Το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιετές 2014-2020 ε, ε, παρουσιάστηκε πέρσι και στις 6 Ιουλίου φέτος ε, υποβλήθηκε μια επικαιροποιημένη έκδοση από την Κομισιόν. Ε, βεβαίως βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο ε, εμπίπτει, καλύπτεται από τις προτάσεις αυτές και βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τελευταία ενημερωμένη έκθεση της Κομισιόν του Ιουλίου. Αυτή η ενημερωμένη επικαιροποιημένη έκθεση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση εργασίας της Επιτροπής που είναι επί της ουσίας και βεβαίως και εμείς πρέπει να ακούσουμε τις απόψεις των άλλων επιτροπών για αυτή την έκθεση. Αυτή η γνωμοδότηση λοιπόν δεν θα καλύπτει θεσμικά θέματα όπως την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξέβρεση συνένεσης και άλλα συναφή θεσμικά θέματα. Η γνωμοδότηση αυτή θα δώσει ένα μήνυμα, ένα σινιάλο ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές δράσεις μέσα στο πλαίσιο της πρόθεσης της ανταγωνιστικότητας και θα απαντά σε γενικές γραμμές ε, στην κατανομή των πιστώσεων και στα συναφή κεφάλαια του προϋπολογισμού για εξωτερικές δράσεις. Επίσης, η ενδιάμεση έκθεση του Κοινοβουλίου θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει τέλος Οκτωβρίου. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή αναγκάστηκε να προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να έχουμε επαρκή χρόνο διαβούλευση και να έχουν και επαρκή χρόνο οι συζητητές. Ε, προτείνει ορισμένα σημεία, αναφέρεται σε ορισμένα σημεία κλειδιά. Το πολιετές χρηματοδημοσιονομικό πλαίσιο δεν αναφέρεται σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Θα πρέπει να μπορέσει να παίξει τον δικό του ρόλο και να τονιστεί ιδιαίτερα λόγω της σημασίας του. Γι' αυτό πρέπει να υπεραμεινθούμε όλων των ε, συμφωνιών που έχουν γίνει μέσα στις, ε, στο πλαίσιο της γυπνίασης και των άλλων συμφωνιών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη των γειτόνων μας ε, και εν ώψη των τελευταίων γεγονότων της Βορείου Αφρικής πρέπει να εξασφαλίσουμε και την υποστήριξη αυτών των εμπορικών μας εταίρων. Βεβαίως, ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα επαρκές, μια, μια ευελιξία, ένα ποσοστό ευελιξίας για την διάθεση των πιστώσεων. Τα έξι αυτά χρόνια, 2014-2020, πιστεύω θα μας δώσουν τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια αυτού του πολιετούς πλαισίου να ανταποκριθούμε με μεγαλύτερη ευελιξία σε κρίσεις, ξαφνικές αλλαγές, ε, δεδομένου ότι ζούμε σε ένα διεθνοποιημένο και μεταλλασσόμενο κόσμο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, που αναφέρατε. Βεβαίως αυτό το MFF, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχει ιδιαίτερη σημασία για τα επόμενα εξι χρόνια, 2014-2020. Δεν αφορά την ουσία ή την αλλαγή στην κατανομή των πιστώσεων, αλλά αφορά την ακρίβεια με την οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι δράσεις τις οποίες καλύπτει και οι οποίες εμπίπτουν μέσα στο πλαίσιο αυτό με τους, ε, τα κατάλληλα ε, κεφάλαια και υποκεφάλαια του προϋπολογισμού έτσι ώστε να μπορέσει να ε, προαχθεί η πρόσβαση στις αγορές. Ε, μήπως υπάρχει κάποιο σχόλιο από τα μέλη μας. Όχι. Ωραία. Ας ακούσουμε την Επιτροπή λοιπόν. Ο κύριος Φόντορκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο επί αυτού του σχεδίου γνωμοδοτήσεως. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με τα σημεία που αναφέρει η συγγητής. απλώ θα ήθελα να πω ότι οι διεθνεί, οι οι συναλλαγές και οι συναφείς στόχοι εμπίπτουν σαφώ στα συγκεκριμένα κεφάλαια εξωτερικών σχέσεων, εξωτερικών δράσεων. Και όσον αφορά την αβεληξία, διάφορες ρυθμίσεις έχουν ήδη εισαχθεί υπό τα ε, διαφορετικά μέσα τα οποία ήδη υπάρχουν στη διάθεσή μας. Υπάρχει λοιπόν το στοιχείο της ευελιξίας. Ο Πρόεδρος, κάποια άλλη παρατήρηση. Ωραία, έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε και τη συζήτησή μας στο σημείο 6 και τροπολογίες είναι ε, προθεσμία την επόμενη Παρασκευή 7 ε, Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, 12 η ώρα. Και Οπότε λοιπόν προχωρήσαμε και έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση των θεμάτων πριν την ψηφοφορία, αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε και το χρονοδιάγραμμα που έχουμε προβλέψει για την ψηφοφορία. Δεν μπορούμε λοιπόν να περάσουμε αμέσω. Πρέπει να κάνουμε μια 15 λεπτή διακοπή.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 Please. Take your seats, please. Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Please conclude your conversations. Take your seats. Let's free... Παρακαλώ αφήστε τις συνομιλίες και καθίστε για να συνεχίσουμε. Oh, what happened? What happened? Excellent. So this is Ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας. Uh, this file, keep quiet. We will vote the... Θα ψηφίσουμε λοιπόν την έκθεση, την γνωμοδότηση μάλλον του κυρίου Πέτερ Στσάσνη ε, για ένα θέμα που, για το οποίο είναι κατ' ουσίαν αρμόδια η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αφορά το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, δηλαδή για το χρόνο. Θα ψηφίσουμε δύο διαφορετικά πράγματα, δηλαδή θα ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες στην γνωμοδότηση που θα κοινοποιήσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και μετά θα ε, ψηφίσουμε τις ε, για τον προϋπολογισμό. Είναι δύο διαφορετικοί κατάλογοι ψηφοφορίας που μας έχει δώσει ο συγγητής μας, ο κύριος Τσάστινη. Πρώτα θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές Ηλεκτρονικό έλεγχο, γιατί δεν προκύπτει με το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την τροπολογία 4. Ο κύριο Κάσπαρ είναι κατά, αλλά ξέχασε την κάρτα του. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται μάλλον. Δεύτερο τμήμα τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, της τροπολογίας 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Adopted. 10 against 9. 10 προς 9. 10 υπέρ, 9 κατά. Τροπολογία έξι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα άρχιτη ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 12. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος ε, για την τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Η τελευταία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Παψήφι εγκρίνεται με 18 ψήφους και μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας για την πρώτη αυτή επιτυχία και περνάμε τώρα στις διάφορες τροπολο... τροπολογίες για τις δημοσιονομικές γραμμές. 69-25, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 69-26, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 69-27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69-28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69-29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69-30. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69-31. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69-32. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και 69-33. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος αλλά ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία δεν χρειάζεται καν ε, τελική ψηφοφορία εγκρίνονται και η γνωμοδότηση και οι τροπολογίες για τον προπολογισμό. Οπότε ολοκληρώνουμε την ψηφοφορία μας και περνάμε στο σημείο 8. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι αν ολοκληρώσουμε την δημόσια μας συνεδρίαση πριν το αναγκαλθέν χρονοδιάγραμμα θα αρχίσουμε αμέσως μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν θα περιμένουμε τις 5.30. Εντάξει. Πολύ ωραία. Προχωράμε στο σημείο 8. Πρόκειται για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για την ε, προσαρμογή των ε, πινάκων σε ό,τι αφορά τις πίνακες δημοκρατίας Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τροποποίηση των παραχωρήσεων. Γιατί οι εξωτερικοί πίνακε γίνονται πιο κοινοτικοί, οπότε θα πρέπει να δοθούν αντισταθμιστικά μέτρα στι Ηνωμένες ε, Πολιτείες για τις υψηλότερες ε, υψηλότερους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχέση με αυτές που εφάρμοζαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Αντίστοιχε περιπτώσεις είχαμε και την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αργεντινή. Πρόκειται για μια κατηγορία συμφωνιών που δεν δημιουργούν προβλήματα. Πρόκειται για εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της ΓΚΑΤ ε, με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 6 ε, ενώπιον της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Γιατί είναι υποφαινόμενος, το θέμα είναι απλούστατο. Το ανέλαβα εγώ για να διεκπαιρεωθεί απλά και εύκολα. Δεν ξέρω αν οι σκιώδεις ηγητές έχουν σχόλια για το σημείο 8. Δεν βλέπω και κανένα σχόλιο από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής μας. Δεν επίβαχο με το θέμα. Δεν ξέρω θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει κάτι. Ο κύριος Βιντσκόφσκι, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω με λίγα λόγια το υπόβαθρο του άρθρου 24.6 και των σχετικών διαπραγματεύσεων. Κάτι λέει εκτός μικροφώνου, δυστυχώς ο Πρόεδρος. Και να σας ε, δώσω μια γενική επισκόπηση της ε, συμφωνίας αυτής. Ό,τι αφορά το ιστορικό υπόβαθρο των διαπραγματεύσεων του άρθρου 24.6. Στόχος μας είναι να συμφωνήσουμε σε μια αμοιβαία ε, ικανοποιητική αντισταθμιστική προσαρμογή ε, μετά την επέκταση της Τελωνιακής Ένωσης στη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Δεν προβλέπονται νέες παραχωρήσεις, αλλά δίνονται αντισταθμιστικά μέτρα στα μέλη του ΠΟΕ για τις απώλειες που υπέστησαν εξαιτία των υψηλότερων δασμών που καλούνται να πληρώσουν σε χώρες που έχουν στο μεταξύ προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Τελωνιακή Ένωση. Αυτό προβλέπουν οι κανόνες του ΓΚΑΤ. Πρόκειται για μια απλή συνηθισμένη διαδικασία, όπως είπε και ο εισηγητής. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε αντίστοιχες συμφωνίες με πολλές χώρες, Κούβα, Βραζιλία, Αργεντινή, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Και μετά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007 έχουμε κρεμίσει δύο συμφωνίες που θα πρέπει να διεκπαιρεώσουμε με την Κίνα αφενός και με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφετέρου. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε, το κείμενο ε, το υποβάλαμε εμείς το Δεκέμβριο και το ε, σχολίασαν τον Φεβράριο οι Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα συζητήθηκε στην Επιτροπή στο σχέδιο ε, του κειμένου πριν την επίσημη έναρξη διαδικασία. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα συστήθηκαν το 2009 και 2010 σε διάφορε τεχνικέ συνεδριάσει και τα βασικά στοιχεία του πακέτου αντισταθμίσεων περιλαμβάνουν καταρχήν μια αύξηση των ποσοστώσεων ε, πουλερικών και γαλοπούλας ε, αύξηση ε, των ποσοστώσεων κατά 200 τόνους στο χείριο κρέας και δημιουργία μιας ποσοστόση. 1515 για παρασκευάσματα τροφών. Τα υπόλοιπα προϊόντα που αναφέρονται στη συμφωνία α, ε, περιλαμβάνονται σε, στη συμφωνία της ΠΟΕ με βάση προηγούμενες ποσοστώσεις ε, των πινάκων Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Επίσης, το άρθρο 2 της συμφωνίας ε, προβλέπεται συμπερίληψη της Ρουμανίας και Βουλγαρίας στις, ε, στις ε, προτινόμενες ποσοστώσεις που θα χορηγήσει η ΕΠΑ ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τυρί. Έχουμε υποβάλει δύο ξεχωριστέ προτάσει για αποφάσει του Συμβουλίου, προκειμένου να διεκπαιρεωθεί η συμφωνία. Η πρώτη ε, επιτρέπει την υπογραφή τη συμφωνία και η δεύτερη οριστικοποιεί τη συμφωνία. Και μάλιστα με την πρόταση εξουσιοδότησης για την ε, σύναψη φωνίας ε, βρισκόμαστε σε προχωρημένο επίπεδο και ζητούμε τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συναυθεί αυτή η συμφωνία πριν ε, λάβει χώρα η υπογραφή της τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Yes. Ωραία. Μας ενδιαφέρει η τάχη στη διεκπαιρέωση του ζητήματος. Εάν λοιπόν και όταν πρέπει να συμφωνήσουμε θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Και έτσι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε πολύ εύκολα επί του θέματος. Θα αποστείλουμε την, το προσχέδιο έκθεσης με μετάφραση μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου εν ώψη της συνεδρίασής μας του Οκτωβρίου. Και στο μεταξύ αναμένουμε την υπογραφή της συμφωνίας από το Συμβούλιο. Άρα το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. 24 Σεπτεμβρίου, αποστολή της έκθεσης και μετάφραση, μετά εξέταση στην Επιτροπή μας στις 10 και 11 Οκτωβρίου, η υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 15 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι και αποστολή τροπολογιών για μετάφραση 17 Οκτωβρίου. Θα ψηφίσουμε ανάλογα με την ε, υπογραφή της συμφωνίας στο Συμβούλιο στις 6 Νοεμβρίου. Και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή. Um, item 9. 9. Συστάσεις προς το Συμβούλιο, Επιτροπή και την Εξωτερική Υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την, για την ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Καζακστάν. Επί της ουσίας θα αποφανθεί η ΑΦΕΤ και εμείς θα γνωμοδοτήσουμε επίσης. Ο δικός μας συγητής είναι ο Μπέρτ Λάγκε. Θα πρέπει να δράσουμε τάχιστα αν θέλουμε να συνεισφέρουμε, διότι η ΑΦΕΤ έχει ένα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα και απέριψε την υπόδειξή μας να παρατείνουμε την προθεσμία. Θα πρέπει λοιπόν να αποφανθούμε. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το γνωστό κανάλι, δηλαδή τη μετάφραση προς τις άλλες γλώσσες εκτός από τα αγγλικά. Οι συντονιστές λοιπόν αποφάσισαν να προχωρήσουμε με αυτούς τους περιορισμούς και γι' αυτό το προσχέδιο θα διατίθεται μόνο στα αγγλικά. Οι τροπολογίες επίσης θα υποβληθούν στα αγγλικά. Αυτό συμφώνησαν οι συντονιστές. Θέλω να το δεχτείτε και εσείς. Δεν υπάρχει λοιπόν αντίρρηση. Δίνω το λόγο στον Μπέρντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Καζακστάν διαβουλεύεται παράλληλα αφενός με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εταιρική συμφωνία και αφετέρου με τον ΠΟΕ για την ε, συμμετοχή, να γίνει μέλος, για να γίνει μέλος. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ένταξη του Καζακστάν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου παρόλο που υπάρχουν ακόμα ορισμένοι τομείς, ορισμένα σημεία στις διαβουλεύσεις που εκκρεμούν. Αλλά η ένταξη ε, του Καζακστάν στον ΠΟΕ νομίζω θα ενισχύσει τη θέση του και γι' αυτό υποστηρίζω την ένταξη του Καζακστάν και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει του χρόνου έτσι ώστε να καλύπτεται από όλους τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις του ΠΟΕ. Το Καζακστάν βεβαίως ενδιαφέρεται σερμά ε, για τις εξαγωγές πρώτων υλών όσον αφορά το πετρέλαιο, όσον αφορά ορυκτά, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, δεδομένου ότι οι εξαγωγές του σε πρώτε ύλες ε, από απόψεως όγκου είναι πολύ μεγαλύτερες από τον όγκο των εξαγωγών άλλων προϊόντων. Γι' αυτό, εάν θέλουμε να έχουμε εμπορικές συναλλαγές, θα πρέπει να μείνουν και ανοιχτές οι θύρες πρόσβασης ε, στις εμπορικές συναλλαγές αυτές. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα στο Καζακστάν, δεδομένου ότι δεν δέχονται τις σεμελιώδεις αρχές του εργασιακού δικαίου βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και επίσης υπάρχει μία ιδιόμορφη σχέση εργοδοτών και εργαζομένων στον πετρελαϊκό τομέα, όπου από τις προφορίες που έχω τουλάχιστον έχουν σημειωθεί 17 θάνατοι στον τομέα αυτό. Επίσης, τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά το περιβάλλον και τις ε, κοινωνικές σχέσεις πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν σεβαστά από το Καζακστάν. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό και γι' αυτό συνέταξα αυτό το ψήφισμα. Πρέπει να μπορέσουμε βεβαίως να συμβαστούμε το χρονοδιάγραμμα της ΑΦΕΤ, αλλά πρέπει να προωθήσουμε, να ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα και προσβλέπω και στις συμπληρώσεις ή στα σχόλια από δική σας πλευράς. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, στα αγγλικά θα είναι το σχέδιο γνωμοδότησης και οι αλλά βεβαίως μπορεί να μιλήσει ο εισηγητής στα γερμανικά και όλη μας η μητρική μας γλώσσα. Ε, και το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη... Α, όχι, είναι η Φρανσίσκα Κέλλερ, τελευταία ομιλήτρια. επί του θέματος. Ε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχασα τις πρώτες δύο προτάσεις που είπατε, αλλά τα άλλα τα παρακολούθησα. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Συμφωνούμε στις γενικές γραμμές. Θα θέλαμε όμως να τονίσουμε ισχυρότερα ορισμένα σημεία αναφέρεται εργασιακές σχέσεις, ανθρώπινα δικαιώματα και εμείς έχουμε αυτές τις πληροφορίες των 18 θανάτων, δηλαδή 18 εργαζόμενοι που σκοτώθηκαν, ε, γεγονό που δεν θα έπρεπε να συμβεί βεβαίως και στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι πρώτες ύλε. Ε, δεν νομίζω ότι αρκεί να πούμε ότι επισημούμε το Καζακστάν να, μας, να προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση στις πρώτες ύλε του, δεδομένου ότι μια εμπορική σχέση είναι πάντοτε διμερής. Ε, πρέπει να εδραιώσουμε ένα μοντέλο που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Ιδίως όταν μιλάμε για πρώτες ύλε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις περιβαλλοντικές ε, πτυχές, την αλλαγή του κλίματος και δεδομένου ότι είμαστε στην Επιτροπή Ήτρα. Μην ξεχνάμε και την ε, ανακύκλωση πρώτων υλών ή το, την πτυχή της ανακύκλωσης όπου μπορεί να εφαρμοστεί. Έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα με την παράγραφο 4 σε σχέση με τα IPR. Είπατε ότι τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εναρμονιστούν. Under review in both και τα δικαιώματα αυτά πνευματικής ιδιοκτησίας ε, πρέπει να συνάδουν με τις αποφάσεις ε, επί του άκτα, τις οποίες έχουμε λάβει εμείς στο σώμα και ή πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη την έκθεση της Κομισιόν για το Καζακστάν που λέει ότι θα πρέπει να, να διευκρινιστούν οι πτυχές της εγχώριας νομοθεσίας σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό επίσης που θα ήθελα να προσέξουμε είναι η ελευθερία πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Καζακστάν που μας ανησυχεί κάπως και όσον αφορά και την έκθεση για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαδίκτυο χωρίς σύνορα. υπάρχουν προβλήματα και στην λειτουργία των διακομιστών του διαδικτύου στο Καζακστάν και ε, έχουν κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διακομιστές μόνο που έχουν την έδρα τους, που λειτουργούν μόνο στο Καζακστάν για τη χρήση του διαδικτύου. Ε, αυτό δεν αφορά μόνο ολόκληρο το ίντερνετ, το διαδίκτυο, αλλά αφορά και την πτυχή της, ε, του ανταγωνισμού. Και ίσως θα πρέπει να αναφερθεί και αυτό στην έκθεση ε, εμείς προς αυτή την κατεύθυνση υποβάλλουμε μία τροπολογία για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε την ε, έκθεσή σας. Αλλά στις γενικές γραμμές συμφωνούμε με αυτά τα οποία λέτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το έργο που επιτέλεσε σε τόσο στενό χρονοδιάγραμμα και ο Πολ Μέρφυ ως και ηγητές ε, ε, κατηγόρησε και εμένα και όλους και ηγητές για το ότι επιβάλαμε τόσο στενόχρονο διάγραμμα στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Πάντως πιστεύω ότι με συνεργασία και κοινέ προσπάθειες θα τα καταφέρουμε. Γενικώ συμφωνώ με τις απόψεις του Μπέρντ Λάγκε. Σε δύο-τρία σημεία μόνο η Γκουε θα υποβάλει προτάσεις για συμπληρώματα. Καταρχήν, ο ρόλος του Καζακστάν είναι σημαντικός. Έχει νευραλγική σημασία στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, που είναι σημαντικός ε, εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα θα πρέπει να θεωρηθεί ως υπόδειγμα στην περιοχή για εργατικά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και από αυτή την άποψη θα πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας ε, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το επισήμανε και η Φραντσίσκα. Και να ε, επικεντρώσουμε την προσοχή μας ε, και στα εργατικά δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα και να υποβάλουμε και σχετικές τροπολογίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το, το νομοσχέδιο και τον εργατικό κώδικα που κατά τη γνώμη συνιστά η παναχώρηση. Και σίγουρα αυτό ο εργατικό κώδικα, η πρόταση εργατικού κώδικα δεν συνάδει με τι διατάξει ε, του Διεθνού Γραφείου Εργασία. Έχουμε και δύο άλλε εκθέσει ε, για το διεθνέ εμπόριο και την εμπορική συνεργασία με τι τρίτε χώρε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτέ τι εκθέσει. Και τώρα θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θα μπορούσε να μας εξηγήσει αν η έκθεση του Ιουνίου του 2012 της Wall Street Journal που ανέφερε ότι μέλη της, ε, μιας επιχείρησης πετρελαίου και μιας ε, γερμανικής εταιρείας έχουν λάβει mail με κατηγορίες για, παράνομη, για παράνομο εκτελονισμό κάποιων προϊόντων. Επίσης υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που δόθηκαν από, το, από τη Wall Street Journal για σχετικές ατασταλίες. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχετικές διευκρινήσεις για τις καταγγελίες αυτές. Και σε ό,τι αφορά το ψήφισμα για το Καζακστάν του ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που ζήτησε, που από την ΕΕΔ να ε, δοθεί συνέχεια στο θέμα της καταστολής της, ε, της διαμαρτυρίας και του συλλαλητηρίου. Τι έχει γίνει από τότε. Και κάτι που ανέφερε η Φραντσέσκα Κέλλερ. Θα υπάρξει ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις α, ε, α, ε, στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Νομίζω ότι στα σημεία αυτά μπορούμε με τα σημεία αυτά μπορούμε να εμπλωτίσουμε την πολύ καλή έκθεση του κυρίου Μπέντ Λάγκη που θα δώσουμε στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ωραία, ολοκληρώνουμε τη συζήτηση και δεν ξέρω αν ε, μπορεί κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Κίθ, να μας δώσει κάποια κάποιες διευκρινήσεις. Δεν κάθομαι στη σωστή θέση και ζητώ συγγνώμη. Βλέπω αντί να κάθεται εκ δεξιών, μου, κάθεται εξεβονίμων η Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να είμαι ουδέτερος ως προς απαντήσεις. Ως προς τα πρώτα ερωτήματα που εθίγησαν, θα ήθελα να πω ότι γενικά συμβαδίζουμε με τα μηνύματα που, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Λάγκε. Μιλάμε για κοινού στόχους σε σχέση με το εμπορικό σκέλος καθώς και το σκέλος επενδύσεων του προσχεδίου. Ε, σε σχέση με την συμμετοχή στον ΠΟΕ, μιλάμε για απότερο στόχο, αυτό είναι απότερο στόχος, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται οι δεσμεύσεις και οι διαπραγματεύσεις. Πολλές φορές υπάρχουν και καθυστερήσεις ως προς διαπραγματεύσεις για ε, ένταξη στον ΠΟΕ και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το εργατικό δίκαιο καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς ε, και συμφωνίες ως προς το πολιτικό σκέλος και την βιώσιμη ανάπτυξη. Σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία και την πλαισίωση καθώς και τις προδιαγραφές έχουν ενταχθεί και στην άκτα Είμαστε σε επαφή με τις αρχές του Καζακστάν για ενημέρωση, για αμοιβαία ενημέρωση. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τους εμπειρογνώμονες που βρίσκονται στην μονάδα προάσπισης ε, πνευματικών δικαιωμάτων να μας πούν πώς εξελίσσεται η συζήτηση. Ήταν ένα από τα τέσσερα κεφάλαια τα οποία συζητήθηκαν κατά τον ε, δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων πριν από τον ε, τρίτο και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συμφωνία αυτή ε, οικονομικής εταιρικής σχέσης. Any further remark? Άλλα σχόλια. Σε σχέση με το άρθρο της Wall Street Journal θα ενημερωθούμε και θα επανέλθουμε επί του θέματος. Εντάξει, ο εισηγητής μας, ο Μπέντ Λάγκε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Είναι πολύ περιορισμένα τα περιθώρια του εισηγητή. Θα πρέπει να εγκριθεί αυτή η πλαισίωση με τροπολογίες βεβαίως και αν θέλετε μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. I explained it at the beginning. Όπως σας είπα και στην αρχή, για τις τροπολογίες έχουμε ορίσει τα, τις προθεσμίες. Θέμα υπαριθμών 10 οι συντονιστές αποφάσισαν στην προηγούμενη συνεδρίαση τους να προετοιμαστεί μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για τα μέτρα για την προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς από εισαγωγές ιδιαίτερα χαμηλού κόστους από την Κίνα, ιδιαίτερα σε αφορά τα φωτοβολταϊκά μηχανήματα και τις τηλεπικοινωνίες. And, uh, I open the floor. Έχετε μπροστά όλα τα στοιχεία στο φάκελό σας και σας δίνω το λόγο. Τι έχετε να πείτε σε σχέση με αυτή την ε, πρωτοβουλία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή αρχή. Βλέπω ότι οι φίλοι μας, οι Γερμανοί έχουν ε, πληγεί ιδιαίτερα. Ο κύριος ε, Λάγκ έχει πρόβλημα με το δάκτυλό του. Ένας άλλος συνάδελφος έσπασε το πόδι του. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό σχετίζεται με την ευρωπαϊκή ανάκαμψη για να ε, επαληθέσουμε την κατάσταση υγείας στην Ευρώπη. Τώρα, πέρα από τους αστεϊσμούς, ως προς τα φωτοβολταϊκά, το συζητήσαμε στους συντονιστές και υπάρχει προφορική ερώτηση και ψήφισμα και πρόταση ψηφίσματος. Ε, αρκετοί συνάδελφοι επανήλθαν στο θέμα της, του ψηφίσματος, άρα παραμένει η προφορική, άλλαξαν γνώμη. Γι' αυτό παραμένει η προφορική ερώτηση κύριος Κασπαρή γνωρίζει ότι μπορούμε να προωθήσουμε τη συζήτηση, αλλά δεν είναι ε, ικανοποιητική για τους οικολόγους, τους οποίους εκπροσωπώ. Μπορούμε να επεκταθούμε και σε θέματα dumping και γι' αυτό ίσως ξεφεύγουμε από την προφορική ερώτηση και υπάρχει ένα θέμα που είναι σημαντικό για μας. Ποια θα είναι επακριβώς η ερώτηση, πώς θα διατυπωθεί. Αφορά την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Δημόσιες Προμήθειες και εάν ναι, ποιες είναι οι, πώς ορίζονται οι γεωγραφικές προτιμήσεις. Μπορεί να μας ενημερώσει η Επιτροπή επί του θέματος. Μιλάμε για μια βιομηχανική στρατηγική η οποία προστατεύει κατά του κινέζικου ντάμπινγκ και αποτελεί και ένα μέσον υποστήριξης για οι επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Πολλές έχουν κλείσει και άλλες γνωρίζουν μεγάλο χρηματοοικονομικό άχθος. Μέχρι αύριο λοιπόν θα πρέπει να υποβληθούν τροπολογίες, όμως οι οικολόγοι θα υποβάλουν ειδικά μία τροπολογία για να τεθεί και το θέμα της γεωγραφικής προτίμησης ιδιαίτερα ως προς τα φωτοβολταϊκά, τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες και ελπίζουμε ότι και οι άλλες ομάδες θα μας υποστηρίξουν. Θα ψηφίσουμε στις 17 ή 18 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια η Ολομέλεια θα αποφανθεί τον Οκτώβριο. <coughs> Ευχαριστώ. Δεν διέφυγε τη προσοχή κανενό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε αντέδρασαν άμεσα και πολύ αυστηρά κατά μιας μεγάλης επιχείρησης dumping ουσιαστικά και αντέδρασαν με επιχορήγηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι μέσα σε λίγα χρόνια οι Κινέζοι κατέκλυσαν ε, όχι μόνο τις ευρωπαϊκές αγορές αλλά και την βορειοαμερικανική αγορά με φωτοβολταϊκούς ε, συλλέκτες σε στα χαμηλές τιμές και μάλιστα 12 κατηγορίες επιχορηγήσεων ε, για παραγωγούς φωτοβολταϊκών συλλεκτών ήταν παράνομη. Αυτό διαπίστωσαν οι ΙΠΑ και μάλιστα οι, παραγωγή, οι Κινέζοι αυτή παραγωγή είχαν τεράστια περιθώρια υποστήριξης 30 ε, με 150% του κόστους ε, του τελικού προϊόντος. Οπότε, εν ονόματι του δικαίου των Ευρωπαίων και των Αμερικανών να υποστηρίξουν ε, τέτοιου βιομηχανίες του μέλλοντος απέναντι σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό εκ μέρους της Κίνας, ε, τέθηκε αυτό το ερώτημα που είναι απόλυτα εύλογο και βάσιμο. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσει και μάλιστα δραστήρια και άμεσα γιατί πρόκειται για μια τεχνολογία του μέλλοντος και μια βιομηχανία του, ε, του μέλλοντος. Δεν μπορούμε να παραγωνιστούμε από την Κίνα και μάλιστα με τέτοιες πρακτικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε και να παρακολουθούμε πολύ στενά την έλαση αυτών των κινέζικων επιχειρήσεων στο, στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Κύριο Σόλτς. Και τώρα ο κύριο από την ΚΟΥΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα, το, το οποίο θίγει και τις διεθνές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και για το μέλλον. Επί της αρχής συμφωνώ και επίσης υποστηρίζω την ε, επέκταση της ε, προθεσμίας αλλά αναρωτιέμαι ακόμα ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι. Άκουσα προσοχή τον Γιάννικ και θέλω να κάνω μια σύνοψη της κατάστασης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα βιομηχανικό τομέα υψηλών ερευνητικών επενδύσεων. Ε, τα φωτοβολταϊκά δεν... Όταν συζητάμε για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, πρέπει να διευκρινίσουμε πού ακριβώς υπάρχουν τα κενά και οι ελλείψεις της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας, του ευρωπαϊκού τομέα και πού προκύπτουν οι μεγάλες ερευνητικές ανάγκες για την ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Στη Γερμανία αυτές οι ευκαιρίες οι οποίες ε, προσφέρθηκαν μετά από την ηλιακή ενέργεια, τις μεγάλες επιδοτήσεις για τις εγκαταστάσεις ηλιακών συλλεκτών, δεν δημιουργήθηκε μία υφόρος προοπτική για το μέλλον όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών και δι των φωτοβολταϊκών. Αν θυμόσαστε είχαν γίνει συζητήσεις επί του θέματος μεταξύ της καγκελαρίου κυρίας Μέρκελ και του Κινέζου ομολόγου. Είχαν πει τότε ότι ας μην προτρέξουμε και προσφύγουμε αμέσως σε ένα διαιτητικό δικαστήριο, ας δούμε καταρχάς πώς εξελίσσεται η υπόθεση και ας δώσουμε νέες προοπτικές στην ευρωπαϊκή, στον ευρωπαϊκό τομέα, στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για να έχει καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη επίσης. Ο Πρόεδρος, υπάρχουν άλλοι ομιλητές? Όχι. Από την Κομισιόν παρακαλώ Ποιος θέλει να μιλήσει, ο κύριος Βέλγε. Α, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ κάθομαι ε, στη διαφορετική θέση σήμερα στην αίθουσα, κάπου στη μέση όμως βρίσκομαι. Κοιτάξτε, έχουμε ε, δυσκολίες στο να αντιδράσουμε και να απαντήσουμε σε αυτό το θέμα. Διότι δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει ε, μία, ένα φάκελο anti-dumping επί του θέματος αυτού που θα ήταν το κατάλληλο μέσο, το κατάλληλο εργαλείο. Από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμευόμαστε να μην δημοσιεύσουμε τίποτα μέχρι ότου ληφθεί η απόφαση εάν θα ανοίξει ο φάκελος προσφυγής ή όχι. Δεσμευόμεθα λοιπόν αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να μιλήσουμε επί της ουσίας. Πρέπει να τηρήσουμε τις νομικές μας δεσμεύσεις και είμαι βέβαιος ότι αυτό το κατανοείτε. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια, το να υποκρινόμαστε ότι τίποτα δεν τρέχει, τίποτα δεν συμβαίνει, είναι πιστεύω πολύ απλοϊκό. Υπάρχουν δεσμεύσεις ε, του ΠΟΕ προς τους συμβαλόμενους και ε, όλους τους εμπλεκόμενους σε, αυτή, σε αυτόν τον τομέα, σε αυτή τη βιομηχανία. Δεν θέλουμε να διακυβευτεί ε, βεβαίως η, βιομηχανία, η βιομηχανία ηλιακών συλλεκτών ή ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανησυχεί ιδιαίτερα εάν τώρα ξεκινήσουμε ένα φάκελο προσφυγής, αν ληφθεί αυτή η υπόφαση, έχουμε 42 μέρες στη διάθεσή μας ώσπου να αποφασίσουμε τελεσίδικα. 42 ε, μέρες από το τέλος του Ιουλίου, σύμφωνα με το ημερολόγιο, με το χρονοδιάγραμμα. Εάν ξεκινήσει αυτή η υπόθεση, και το αποφασίσουμε, θα έχουμε εν συνεχεία 9 μήνες στη διάθεσή μας για προσωρινά μέτρα και γενικά μέσα σε 15 μήνε θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια οριστική απόφαση. Αυτό είναι γενικά το χρονοδιάγραμμα το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε και αυτό μπορώ να σας πω τώρα. Υποθέτω ότι εάν οι συνθήκε συνεχιστούν, αν η κατάσταση συνεχιστεί έτσι, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τις ουσίες του προβλήματος σύντομα. Well, I understand. Ο Πρόεδρος, ναι, κατανοώ ότι η Κομισιόν δεν μπορεί δημόσια να εκφραστεί πριν ληφθεί μία απόφαση αν θα ανοίξει η υπόθεση, η φάκελος επί της υποθέσεως ή όχι. Αλλά ε, από ό,τι ε, ξέρω μπορεί η Κομισιόν ήδη να έχει καταλήξει σε ορισμένε αποφάσεις, ίσως και κλεισμένων των θυρών. Γι' αυτό θα θέλαμε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, ελπίζω να το μάθουμε σύντομα. Τώρα, ε, επανέρχομαι στις εργασίες της Επιτροπής μας. Υπάρχει μια πρόταση να αλλάξει η προθεσμία των κατάθεσης τροπολογιών. Είναι επίσημη πρόταση αυτή να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα. Ο, ο κύριος Υπάρχει επίσημη πρόταση να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Λάγκερ. Προτείνω να γίνει, η προθεσμία να γίνει 8 Σεπτεμβρίου. 8 Σεπτεμβρίου. Α, δηλαδή ανατρέπουμε την απόφαση των συντονιστών, η οποία λήφθη εν τη μου. Οι συντονιστές αποφάσισαν να υιοθετήσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα ώστε η απόφαση να ληφθεί τον Ιανουάριο μετά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Αλλά έχουμε και την απόφαση της Ολομέλειας. Συμφωνείτε με τις επιπτώσεις αυτής της αλλαγής της προθεσμίας. Είναι τόσο σημαντικό να έχουμε μερικές μέρες περισσότερο για τις τροπολογίες ή ήδη είναι πιο σημαντικό να ληφθεί η απόφαση στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Εάν συμφωνείτε ότι είναι καλύτερα να ληφθεί η απόφαση στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου, πρέπει να σεβαστούμε το υπάρχον χρονοδιάγραμμα. Εγώ σας προειδοποίησα για τις επιπτώσεις αλλαγής του χρονοδιαγράμματος. Εγώ πιστεύω ότι πολύ σοφά αποφάσισαν οι συντονιστές για αυτό το χρονοδιάγραμμα που έχουμε τώρα. Υπάρχει τώρα όμως, υπάρχει, εμένεται στην διαφορετική συναλλαγή. Διάλογος εκτός μικροφώνου. Ο πρόεδρος λέει ότι αυτή η υπόψη που έχει ληφθεί είναι πάρα πολύ σοφή, πολύ συνετή και δεν θα αλλάξουμε. Γι' αυτό η τροπολογία, η λήξη δηλαδή της προθεσμίας είναι αύριο, 4 Σεπτεμβρίου. Δεν αλλάζει τίποτα από αυτού. Δεν υπάρχει εισηγητής και εγώ ως πρόεδρος είμαι υπεύθυνο. Υπάρχουν αυστηρές, αυστηρά όρια όσον αφορά στην έκταση των προφορικών ερωτήσεων. Αυστηρά όρια. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό λέξεων. Γι' αυτό σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη τα όρια αυτά και να αντισταθμίσετε τις υποχρεώσεις αυτές ως προς την έκταση των προφορικών ερωτήσεων. Διαφορετικά για ε, τυπικούς ε, λόγους ε, δεν θα δεχτούμε τις τροπολογίες οι οποίες δεν κάνουν σεβαστά αυτά τα κριτήρια. Λοιπόν, μετράτε τις λέξεις παρακαλώ, μετράτε τις λέξεις. Και παρακαλώ να τη συντάξετε με το βέλτιστο τρόπο. Λοιπόν, ανέφερα ήδη το χρονοδιάγραμμα, δεν αλλάζει, άρα λοιπόν ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας, τις εργασίες της ίντα και όποιος δεν είναι ε, μέλος ε, το, της ομάδας των συντονιστών που θα συνεδριάσει τώρα, παρακαλώ να εξέλθει της αίθουσας. Let me remind Να σας θυμίσω, για τους συντονιστές για τη συνεδρίαση των συντονιστών είναι μόνο οι συντονιστές, ο γραμματέας της Επιτροπής, η νομική υπηρεσία, εξηματούχοι των πολιτικών ή εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και όλοι οι άλλοι παρακαλώ να εξέλθουν της αίθουσας. And Και η βοηθή. Όλοι οι άλλοι παρακαλώ ε, να φύγετε από την αίθουσα.